Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την υποστήριξή του γενικά στις προτινόμενες μεταφορές πιστώσεων. Έχουν σημειώσει δύο ερωτήσεις προς εμάς. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Η ερώτηση πρώτη έχει να κάνει με το 19, αυτό το αίτημα μεταφοράς πιστώσεων, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μεταφερθούν 20 εκατομμύρια από υποχρεώσεις για μισθούς για να ενισχυθούν τα συστήματα πληροφορικής. Ρώτησε ο εισηγητή για ποιο λόγο αυτό δεν είχε συμπεριληφθεί στο αρχικό σχέδιο του προπολογισμού στην πρότασή μας. Η βασική εξήγηση είναι ότι οι ανάγκες αυτές προέκυψαν από την πρόσφατα σε ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα τέλη του 2018. Αυτές οι ανάγκες λοιπόν δεν είχαν ακόμα ταυτοποιηθεί ε, ω τέτοιε όταν εγκρίθηκε το σχέδιο του προπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι την Άνοιξη. Αυτό δεν είναι όμως 100% της υπόθεσης, όπως μπορείτε να φανταστείτε ορισμένες από τις ανάγκες αυτές ήταν ήδη γνωστές και ιδιαίτερα εκείνες που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες και απαιτήσει του νέου λογιστικού συστήματος, το σύστημα ΣΟΥΜΑ που έρχεται να αντικαταστήσει το τρέχον ΑΠΑΚ όπως προτείνει ο εισηγητής, εκεί πραγματικά εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουμε κάποιο περιθώριο που υπάρχει στην κατηγορία ε, έτσι ώστε να προωθηθούν αυτές οι αναλήψεις υποχρεώσεων. Αλλιώς θα καλυφθούν μόνο το 2020, αλλά είναι ένα σχέδιο προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαιρόμαστε πολύ που βρήκαμε κάποιο περιθώριο για να καλυφθούν ε, τα έξοδα αυτά το 2019 και ζητούμε την υποστήριξή σα. Το άλλο που ρώτησε ο εισηγητή έχει να κάνει με τη μεταφορά DEC 11, που είναι η ενίσχυση της διαχείρισης κρίσεων, κεφάλαιο 19-1903 για να διευκρινίσω. Οι περισσότερες από τις μεταφορές αυτές ε, αφορά ανάληψη υποχρεώσεων, αλλά αυτό που ρωτάει ο εισηγητής είναι πίστοση πληρωμών. γιατί έχει μεταφορά, το συγκεκριμένο αυτό που ρωτάει στοιχείο. δεν έχει προσμειωθεί για κάποια ειδική χρηματοδότηση είναι ε, αποτέλεσμα Γενικής Εκτίμησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις ανάγκες πληρωμών για το τρέχον έτος. Για όλες τις αποστολές στην ε, κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας και άμυνας. 16 εκατομμύρια πληρωμές θα χρειαστούν. Γι' αυτό ζητήσαμε να ενισχυθεί αυτός ο κλάδος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις έχετε, σχόλια, παρακαλώ. Ο κύριο Ανδρίασεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε ικανοποιημένοι σχεδόν με όλες αυτές τις προτάσεις. Θέλουμε αναβολή της ψηφοφορίας για το ΤΕΚ 15. Εάν δεν μπορούμε να αναβάλουμε, να εξηγήσω γιατί έχουμε πρόβλημα. Σαν πράσινοι θα καταψηφίσουμε αν γίνει ψηφοφορία. Είχαμε εκλογές στην Ελλάδα προ κάποιων εβδομάδων και ο νέος Πρωθυπουργός της Ελλάδας έκανε ε, αναφέρθηκε στα δικαιώματα των προσφύγων και ανέφερε σχέδια να χτίσει κλειστά κέντρα κράτησης για ετούντες άσυλο. Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Κάποια ευρωπαϊκά χρήματα που θα ψηφίσουμε να καταβληθούν, συμμοποιηθούν για να χτιστούν αυτά τα κέντρα. Αυτό μας προβληματίζει. Γι' αυτό προβληματιζόμαστε με αυτή την πρόταση. Χρειαζόμαστε περισσότερε πληροφορίε. Ξέρω ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών αργότερα σήμερα ή αύριο θα συζητήσει το θέμα στην Επιτροπή. Είναι ειδική αυτή στην Επιτροπή αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να τους ακούσουμε. Αν αυτό είναι ανέφικτο για λόγους τεχνικούς, για λόγους προϋπολογισμού, τότε η ομάδα μας θα καταψηφίσει σήμερα. Και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μία μοναδική, μία ενιαία ψηφοφορία αυτό το θέμα και μετά ψηφίσουμε τα υπόλοιπα. Ξεχωριστά αυτό. Δυστυχώ, Δεν ε, έχουμε ε, τέτοιο χρόνο. Ε, υπάρχει πρόβλημα για την αναβολή με το χρονοδιάγραμμα. Αν συμφωνεί ο κύριος Χάουαρτ, θα πρότεινα να ψηφίσουμε το 6 με 14 unblock, δηλαδή μαζί όλες τις μεταφορές και τη 15 ξεχωριστά. Συμφωνείτε κύριε Χάουαρτ, μάλιστα. Πράγματι, ναι. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, μία δοκιμή πρώτα, μία δοκιμαστική ψηφοφορία για να δοκιμάσουμε τα μηχανήματα. Είστε όλοι έτοιμοι. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ε, ε, λείπουν εννέα ε, βουλευτές. Ποιος κρύβεται. Ψηφίζουν εννέα λιγότεροι από όσους θα όφυλαν. Okay. Then we... Είμαστε εντάξει, πέρας λοιπόν της ψηφοφορίας. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν λειτουργεί εδώ το μηχάνημα. Μπορεί να ψηφίσει διανατάσσεως χειρός. Δεν δουλεύει το μηχάνημα. Those have machines, please vote. Παρακαλώ ψηφίστε όσοι έχετε τα μηχανήματά σας που λειτουργούν. It's not working. Okay, then uh, I propose that we... Καλώς. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά όσοι μπορούμε και οι υπόλοιποι διανατάσεως της χειρός όταν δεν λειτουργούν τα μηχανήματα. Είμαστε έτοιμοι. Ψηφίζουμε λοιπόν το DEC 6 μέχρι και DEC 14. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote, is closed. Πέρασε. ψηφίζουν, 28 υπέρ, 3 αποχές και 5 κατά. So, οι μεταφορέ αυτές εγκρίνονται λοιπόν DEC 6 μέχρι και DEC 14. Τώρα θα ξαναψηφίσουμε ξεχωριστά την DEC 15 παρακαλώ. Άρχεται η Ψηφίσατε όλοι. Περάσε. And DEC 15 is also adopted. Εγκρίνεται και η μεταφορά DEC 15. 25 υπέρ από 36 σύνολο ψηφισάντων. This closes our point 12 on σημείο 12 λοιπόν φτάνουμε στην μοίραση δίταξη. μάλλον το τελειώσαμε και πάμε στο 13 και θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Φερνάντες για να μας παρουσιάσει τις μεταφορές πιστάσεων και τις τροποποιήσεις ε, των, ε, της κατάστασης ε, προβλέψεων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές οι αλλαγές είναι ουδέτερες για τον προπολογισμό. Συνεπώς δεν έχουμε νέα ποσά. Πρόκειται περί μεταφορών σύμφωνα και με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μάλλον για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πρόκειται για το κονδύλιο, παλιό κονδύλιο 1400, άλλοι απασχολούμενοι. Εκεί προβλέπονται 750.000 για την κάλυψη έξι συνεργατών που πρόκειται να προσληφθούν στο δεύτερο εξάμεινο του έτους. Πάλι για το οργανόγραμμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόκειται για ένα κονδύλιο 80.000 ευρώ για, την, για να αντιμετωπιστούν αυξήσεις μισθών άλλα κονδύλια προβλέπονται για την προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Κονδύλιο 14-19 αύξηση κατά 200.000 ευρώ. Αυτό πρόκειται να καλύψει ανάγκες που έχουν προβλεφθεί από την αρχή του έτους και για το 14.016, 14.06 μάλλον, 14.000 ευρώ για την παράταση συμβάσεως εργασίας ενός συνεργάτη στην, ε, στο τμήμα ορκωτών λογιστών, στο τμήμα δηλαδή ε, ε, οικονομικών ελέγχων. Παρακάτω 100.000 ευρώ στο κονδύλιο 14630 για μεταφράσεις δημοσιεύσεων και νέων δημοσιεύσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την διευκόλυνση της εργασίας δημοσιότητας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόκειται λοιπόν για μεταφορά πιστώσεων για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, άλλο κονδύλιο για την αύξηση για την αντιμετώπιση δαπανών ε, εστιατορίων για την αγορά για την αγορά σκευών ε, από άλλες ύλες εκτός πλαστικού. 300.000 ευρώ προβλέπονται για το κονδύλι αυτό, από τις οποίες 30.000 για την ανακύκλωση των μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενων σκευών. Άλλες μεταφορές κονδυλίων για τον καθαρισμό και συντήρηση του κτηρίου 17.000 ευρώ για εργασίες συντηρήσεως και για την παράταση των σχετικών συμβάσεων άλλες μεταφορές πιστώσεων πάντα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 8.019 2318, αύξηση κατά 10.000 ευρώ. Πρόκειται για έξοδα μετακόμισης γραφείων από το κτίριο K2, το οποίο πρόκειται να ανακαινιστεί το φθινόπωρο. Στην διάρκεια δηλαδή των εργασιών ανακαινήσεως, οι συνεργάτες θα στεγαστούν σε άλλο κτίριο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπάρχει κι άλλη μια μεταφορά πιστώσεως Α19 για την αύξηση για ηματισμό εργασίας. Ιδίως διότι πρόκειται να προσληφθούν νέοι υπάλληλοι στην ασφάλεια του κτηρίου και γι' αυτό έχει ζητήσει αύξηση του κονδυλίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και πρόκειται για 1.000 ευρώ στο κονδύλιο 1220, 1220. Επίσης το VAB Α19 και το κονδύλιο 2770 τεκμηρίωση, βιβλιοθήκη και αρχείο Προβλέπετε ποσό 25.000 ευρώ έξτρα δαπάνες για τη συντήρηση του ιστορικού αρχείου και για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του αρχείου αυτού. Επίσης για τη μεταφορά VAB 12 c 19 80.000 ευρώ για τον καλύτερο εξοπλισμό του ιατρικού κέντρου. Άλλο κονδύλιο για, για το οργανόγραμμα. Εδώ κατ' εφαρμογή του άρθρου 53 του κανονισμού. όπου μία θέση διοικητικού υπαλλήλου θα χωριστεί σε δύο θέσεις τύπου ADS μετά από την αποχώρηση δύο συνεργατών AST. Και τελευταία ε, μεταφορά πιστώσεως ήταν αυτή τώρα του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Τώρα ερχόμαστε στην Επιτροπή Περιφερειών στον τίτλο 214 για τη συντήρηση αιθουσών του κτηρίου. Οργανόγραμμα τώρα του ίδιου οργάνου, Επιτροπής Περιφερειών. Πάλι κατ' εφαρμογή του άρθρου 53 του κανονισμού για προσωρινή σύμβαση εργασίας AD6 και για να μετασχηματιστεί θέση προσωρινού υπαλλήλου σε μόνιμο. Αυτά για την ε, Επιτροπή Περιφερειών και τέλος έχουμε το γραφείο του εντεταλμένου την προστασία προσωπικών δεδομένων που προτείνει μεταφορά πιστώσεων 550.000 ευρώ για αναγκαίες προσλήψεις. Χρειάζεται δηλαδή εκεί να συναυθούν συμβάσεις εργασίας. Και για τον συνήγορο του πολίτη πάντοτε κατ' εφαρμογή του άτου 53 του κανονισμού. Πρόκειται για πρόσληψη εργαζομένου ASD4. αναγκαίος σχεδιασμός δηλαδή για την διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων. Εγώ πάντως προτείνω έγκριση των ε, προτινόμενων μεταφορών πιστώσεων. Εάν βέβαια υπάρχουν ε, περαιτέρω ερωτήσεις, υπάρχουν εδώ παρόντες εκπρόσωποι των ε, διαφόρων αυτών οργανισμών που μπορούν να δεχθούν ερωτήσεις. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Φερνάντες. Έχετε σχόλια ή ερωτήσεις. Η κυρία Γουάρτια Ζαμπάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι. Εμείς θα υπερψηφίσουμε όλες τις μεταφορές πιστώσεων, αλλά είχα ένα διευκρινιστικό ερώτημα, έτσι, ενημερωτικό για το ελεκτικό συνέδριο για τη μεταφορά πιστώσεων για την ιατρική υπηρεσία. Από ό,τι κατάλαβα είναι για να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις και να αυξηθεί η ε, ικανότητά τους. Γιατί έχει αυξηθεί η ζήτηση τώρα προς την ιατρική υπηρεσία. Υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος. Κατανοώ ότι μπορεί να είναι ευαίσθητες αυτές οι πληροφορίες και εμπιστευτικές και να μην δηλώνονται δημόσια γιατί πρόκειται για την ιατρική υπηρεσία. Αλλά θα μου φαινόταν ενδιαφέρον. Είπα θα υπερψηφίσουμε τη μεταφορά πιστώσεων, απλώ με ενδιαφέρει για ποιο λόγο έχουν αυξηθεί οι ανάγκε και η ζήτηση τη ιατρική υπηρεσία. Αν δεν μπορείτε να μα το πείτε εδώ, να μα το διαβιβάσετε με τον τρόπο που εσεί φρονείτε σκόπιμο. Thank Ευχαριστώ. Έχετε άλλα σχόλια. Εάν όχι, τότε για το ερώτημα τη κυρία Γουάρια θα δώσω το λόγο στον κύριο Φέντε την κυρία μάλλον, ε, το, η ιατρική υπηρεσία του ελεγκτικού συνεδρίου κάνει συντήρηση των εγκαταστάσεων, διότι για την ώρα έχει μόνο δύο μικρές αίθουσες. Επειδή λοιπόν προσελήφθησαν τώρα νέοι εργαζόμενοι, είχαμε πολλές καινές θέσεις, τώρα έχουμε λίστες από καταλόγους δηλαδή από διαγωνισμούς και προσλαμβάνουμε ανθρώπους και αυτοί βέβαια πρέπει να περάσουν τις ιατρικές τους εξετάσεις. Γίνονται επίσης οι έλεγχοι των οδηγών και επομένως υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση των υπηρεσιών του, της ιατρικής υπηρεσίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι νοσεί περισσότερος κόσμος, ότι υπάρχουν σημειώνονται περισσότερες ασθένειες, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, φτιάχνουν του φακέλου του και προσλαμβάνονται κτλ. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Άλλα σχόλια ή ερωτήσει. Όπω λοιπόν εξήγησε προηγουμένω ο κ. Φερνάντε, δεν βλέπω και εγώ να υπάρχουν ενστάσει. Επομένω, οι μεταφορέ πιστώσεων για το οργανόγραμμα εγκρίνονται. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Τώρα το υπαριθμόν 15 πολιτική ακινήτων. Δυστυχώς οι συντονιστές δεν αποφάσισαν ακόμα για το ποιο μέλος τους θα αναλάβει την ευθύνη των ε, σχετικών φακέλων, άρα θα πρέπει να δεχθείτε να κάνω εγώ την ε, ε, πρόταση για το EES η Υπηρεσία δηλαδή Εξωτερικών Δράσεων που προτείνει να ε, κάνει μια μακρόχρονη μίσθωση ε, για τη κτηρίου στην Ιανγκόνγκ της Μιανμάρ για να έχει δηλαδή να βρίσκεται τα γραφεία της σε κατάλληλη ε, τοποθεσία. Αυτό έχει δοθεί ως έγκαιρη προειδοποίηση στην διάρκεια βέβαια του, της διακοπής για τον προεκλογικό αγώνα τα κτίρια που υφίστανται τώρα είναι βέβαια σε καλή κατάσταση, αλλά είναι της ποιότητας και έχουν πολλά προβλήματα ασφαλείας και κυρίως ε, σε ό,τι αφορά την αντοχή τους σε σεισμούς. Υπάρχουν άλλα κτίρια λοιπόν υποκατασκευή εκεί κοντά. Προτείνεται λοιπόν αλλαγή του κτιρίου με καλύτερε αντισυσμικέ προδιαγραφέ, καλύτερη λειτουργικότητα και καλύτερη αποδοτικότητα χρήση ενέργεια και καλύτερη ορατότητα από αυτά που έχουν τώρα. Το συνολικό κόστος των νέων κτίριων, θα σας πω τα νούμερα, θα είναι περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ για 10 χρόνια. Και σε αυτά περιλαμβάνονται και το κόστος λειτουργίας και ε, συντήρησης. Και θα συστεγαστούν με άλλους οργανισμούς. Σύμφωνα με το αρχικό σημείωμα της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων, επρόκειτο να συστεγαστεί με την Πολωνική και Ισπανική Πρεσβεία καθώς και με τον οργανισμό ΕΚΟ. Χθες όμως η υπηρεσία μας, μας ειδοποίησε χθες ότι δεν θα συμμετάσχει η Πολωνία, άρα θα υπάρξει κάπως υψηλότερο κόστος. Τη τάξη δηλαδή η διαφορά θα είναι των 400.000 ευρώ. Το καθαρό κόστος της παραμονής στα παρόντα κτίρια θα ήταν 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο, Κάτι ξέχασα πριν. Η προσωπία εξέτασε και το ενδεχόμενο ε, να προβεί σε αγορά. Όμως, νομικά είναι αδύνατον, δεν επιτρέπει δηλαδή η ε, νομοθεσία της ε, Μπούρμα να αγοράσουν μη Βυρμάνοι μη έχονται στην εθνικότητα ακίνητα στην περιοχή αυτή. Βεβαίω, επισημαίνουμε στου εκπροσώπου τη ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων την υποχρέωσή του να ενημερώνουν πλήρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με κάθε βήμα που κάνουν. Τώρα, θα παρακαλέσω τον κύριο, την κυρία μάλλον Βάσκεθ ε, τη Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων να ενημερώσει την Επιτροπή Προπολογισμών. Σα ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στους βασικούς λόγους για την πρόταση μετακίνησης. Όπως είπατε, είναι απαραίτητες οι βελτιώσεις από πλευράς ασφαλείας και αντοχής του κτηρίου. Από την αρχή, όταν η αντιπροσωπή εξέτασε τη δυνατότητα της μετακόμισης, Βασική μας μέρημνα ήταν και η οικονομική δυνατότητα. Τα κίνητα στη Μιανγκόγκ γινόταν όλο και πιο φθηνά. Οπότε τότε θα γλιτώναμε 30-40% από τις μειώσεις των τιμών. Αυτό που συνέβη στο μεταξύ και το βλέπετε στους πίνακες ότι έπρεπε να παραταθεί τον Απρίλιο για ένα χρόνο η μίσθωση για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες που συζητούμε. Όταν ανεώθηκε η μίσθωση τον περασμένο Απρίλιο, ο ιδιοκτήτης έκανε επιθετική πρόταση, μείωσε την τιμή κατά 30%. Άρα συγκριτικά έρχεται περίπου ε, ίδια είναι η κατάσταση οικονομική. Η διαφορά είναι τόσο σημαντική όσον αφορά τιμή όπως στην αρχή. Ακόμα και αν είχαμε, δεν είχαμε καμία μεταβολή. Έχουμε όμως καλύτερη ασφάλεια, ε, αξιοπιστία του κτηρίου, καλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, πιο ποιοτικό κτίριο. Διότι εμείς των τιμών στην περιοχή ε, οδήγησε και στην βελτίωση των κτηρίων, την ποιότητα των κτηρίων. Οπότε, αναφερθήκατε στο δυνατότητα αγοράς Υπάρχει και θέμα πολιτικό. Πολιτική ευκαιρία παρουσιάζεται. Όπως ξέρετε, η διοικητική πρωτεύουσα του Μιανμάρ έχει μετακινηθεί. Έχει, έχει πάει στο Ναπιτάο. να Ενθαρρύνουν οι αρχές τις διπλωματικές αποστολές να μετακομίσουν, να πάνε στο Ναπιτάο. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί διότι δεν υπάρχουν όλες οι δυνατότητες στην Απιτάο. Κανένα κάτος μέλος δεν πήγε στον Απιτάο. Αλλά πιθανότατα αυτό είναι κάτι που θα γίνει την επόμενη δεκαετία. Εν τη αυτή περιπτώση θεωρήσαμε ότι η αγορά δεν ήταν οικονομικά επωφελής για την Ένωση. Αυτά μπορώ να πω για την ώρα. Ίσως Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, διότι έπρεπε να είχαμε στείλει χθε επικαιροποιημένο οικονομικό πίνακα χθε. Μόλι τη Δευτέρα μάθαμε όμω ότι η Πολωνία, την περασμένη Παρασκευή, ότι η Πολωνία θα αποσυρθεί από το πρόγραμμα. Ε, Ευτυχώ η πολωνική συμμετοχή ήταν πολύ μικρή, δύο γραφεία. Ένα ενάμιση όροφο είχε. 2,5% από πλευράς έκτασης και από πλευράς οικονομικής Άρα δεν κάνει τη μεγάλη διαφορά, κατά την άποψή μας, όσον αφορά το θέμα που εξετάζεται. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν σχόλια, υπάρχουν ερωτήσεις από τους παρισταμένους. Αν δεν υπάρχουν, προτείνω να ψηφίσουμε αυτό το θέμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται η πρόταση 27 με 36. 27 ψηφί. Πέρα τους 36 ψηφίσαντε, συγγνώμη. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία μας. Πάμε στο σημείο 16 ημερησίας διάταξης, ετήσια συνάντηση με τους διάφορους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διάφορες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτό των σχέσεων στα πλαίσια του ετησίου προπολογισμού με τις υπηρεσίες. Για τον σχέδιο προπολογισμού για το 2020, για τα νέα μέλη, να πω ότι θα ήταν σκόπιμο να μάθετε το σκοπό και τη λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία από πλευρά δημοσιονομική. Γι' αυτό αυτή η ανταλλαγή απόψεων σημερινή μπορεί να αναφερθεί και σε γενικότερες πτυχέ πέρα από τις τροποποίησεις του δύο προπολογισμού για το 2020. Θα έχουμε ομιλητές την κυρία Μον, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη των Ασθενειών, είναι εδώ από την ιδιότητά τη ω ο παρούσα πρόεδρος της, του δικτύου ε, της υπηρεσίας αυτής, της Τρόικα. Η κυρία Ντεμπόλα επίσης, εκτελεστική διευθύντρια της Europol και είναι και ο κύριος Μαρτίνο, υποδιευθυντής για θέματα διοίκηση. Τέλος, ο κύριος Κι Ικάη, εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών. Η πρόταση για μόνιμο εισηγητή για τις υπηρεσίες εκκρεμεί. Ο προϋπολογισμός για το 2020 είναι κάτι που θα παρουσιάσει η κυρία Χολμάιερ για αυτή τη φορά. Έχετε το λόγο. Που είναι εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και τους οργανισμούς, ευθύς εξ αρχής θέλω να πω ότι αναλαμβάνουν αυτοί οι οργανισμοί κάποια καθήκοντα ε, που προκύπτουν και από την εκτελεστική εξουσία ε, και που τα τελευταία χρόνια έχουν ε, αναγκαστικά διευρυνθεί, γιατί έχουν αυξηθεί και οι αποστολές και τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ε, ένα ε, εισόδημα από τέλη που ε, συλλέγουν οι οργανισμοί και μάλιστα συνιστούν ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων τους για πολλούς οργανισμούς και έτσι ελαφρύνεται σημαντικά ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ωστόσο, ως Επιτροπή Προϋπολογισμών εμείς ανέκαθεν λέγαμε ότι οι αρμοδιότητες που πρέπει ε, να ε, ε, είναι στα χέρια του δημοσίου θα πρέπει να χρηματοδοτούνται και από το δημόσιο. Αλλιώς έχουμε προβλήματα σύγκρουση συμφερόντων ή και λειτουργίας των οργανισμών. Γι' αυτό χαίρομαι που έχουν έρθει εκπρόσωποι των οργανισμών. Ευχαριστώ για την επικοδομητική συνεργασία που ανέκαθεν είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί σας. Στο σχέδιο προπολογισμού τώρα για το έτος 2020 όλοι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί θα πρέπει ε, να χρηματοδοτούνται με ένα ποσό της τάξης των 1,777 δισεκατομμυρίων. Έχουν ήδη εγγραφεί ε, οι ε, δαπάνες αυτές μαζί με τα έσοδα και υπάρχει και ένα πλεόνασμα από το 2018, 38,6 εκατομμύρια. Οι συνολικές δαπάνες των οργανισμών έχουν αυξηθεί σε σχέση με τον προπολογισμό του 2019 ε, ε, κατά 9,7%. Αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τη μετανάστευση και την ασφάλεια και κυρίως με τις αλλαγές που έγιναν στο Frontex. Η αντίστοιχη νομοθεσία εγκρίθηκε στο τέλος της ε, προηγούμενης θητείας και αλλαγές αρχίζουν τώρα από το 2020 και είναι αισθητέ. Ε, η συνεισφορά της Ένωσης αυξάνεται σε σχέση με το 19 κατά 107,3 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν οργανισμοί όπως ο ΕΑΣΟ για το άσυλο που έχει μεγάλη αύξηση 42,1 εκατομμύρια και το ίδιο Λάιζα ε, μείωση 55,6 εκατομμύρια ευρώ που είναι κρίσιμο για μένα και αμφισβητώ πάρα πολύ αυτό το ποσό γιατί έτσι και αλλιώς αυτή, αυτός ο οργανισμός δεν λειτουργεί ε, ως τα όφιλε και θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται. Γιατί τις θεωρούν από παιδιά αυτές τις υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτούς τους οργανισμούς, τους αποκεντρωμένους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και ε, έχουν σημαντικές περικοπές και προβλήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους στην Ευρωπόλ και τα κράτη-μέλη έχουν κάποια αιτήματα τα οποία δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, στο οργανόγραμμα για το 2020 σε όλους τους ε, οργανισμούς έχουμε 7.578 υπαλλήλους και εκεί είναι βέβαια και το άσυλο και η μετανάστευση. 190 επιπλέον, 191 ε, θέσεις ε, για τη Frontex, 125 πέφτουν στη νέα θητεία για τη δημιουργία ε, ενός σώματος σταθερού 10.000 υπαλλήλου, 82 επιπλέον θέσεις για τον οργανισμό ΕΑΣΟ και 20 θέσεις για το EU LISA. Συνολικά έχουμε αύξηση κατά 293 θέσεις ε, το σχέδιο προπολογισμού του 2020 ε, περιλαμβάνει και δύο νέους οργανισμούς που βρίσκονται ακόμα στην ανακτήρια φάση. Το ένα είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέω προσεκτικά ότι έχει αρχίσει με κάποια φιδωλή ε, στελέχωση και, και δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κανείς να στήσει ολόκληρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σοβαρή με τέσσερα πρόσωπα ε, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας επίσης είναι μια καινούργια δομή που ε, ξεκινάει τώρα. Επίσης σημαντικό είναι να έχουμε ε, και την μεσοπρόθεσμη εικόνα στο μυαλό μας, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι από το 2021 μέχρι το 2027 και οι νέοι οργανισμοί ε, θα πρέπει ε, το 2020 να έχουν κάποια σχετικά λογική χρηματοδότηση. Υπάρχουν οργανισμοί που έχουν τεράστια προβλήματα. Ε, ο προπολογισμό και το σχέδιο του για το 2020 θεωρείται από εμά βάση για την έναρξη και όχι το έτος 2018, ναι, το έτος αναφοράς. Αν θέλετε να σας απαντήσω σε λεπτομέρειες στη συνέχεια στη συζήτηση, πάντως με τους οργανισμούς θα πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ εντατικά Ιδιαίτερα επειδή έχω παρακολουθήσει κάποιους φακέλους με θέματα ασφαλείας, ε, υπάρχουν ελλείμματα. Και αν μπορεί, ε, νομίζει κανείς ότι έτσι με μια μόνο κοντιλιά μπορεί να ε, περικόψει 35% των θέσεων του οργανογράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πραγματικά αναρωτιέμαι πώς γίνεται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε εκεί στις αποφάσεις ε, καλά, μπορούμε να τα ρίξουμε ε, στη διοικητική λειτουργία, στη νομική λειτουργία, αλλά αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη μείωση της δυνατότητα συνεργασίας των κρατών μελών και δεν απαντούν και τις ερωτήσεις. Και έχω ρωτήσει τα κράτη-μέλη για να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μέχρι και μία τριετία ε, και προσεχώς πενταετία. Οπότε τι να την κάνουμε την υπηρεσία και τις δυνατότητες και το, την πληροφορική και το προσωπικό αφού δεν απαντάνε στις ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε στις λεπτομέρειες ε, επί της ουσίας και για την εισαγγελία παραλαμβάνω νομίζω είναι ελληματική η στελέχωση. Εάν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να γίνει αυτό που φανταστήκαμε ότι θέλουμε για να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να μπορεί κάπως να λειτουργεί αυτή η δομή. Ε, πράγμα που δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα πετυχημένο με τη σημερινή στελέχωση. Ε, Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οργανισμοί που θα υπάρχουν ε, ε, προβλήματα. Χαίρομαι που έχουν έρθει κάποιοι οργανισμοί για να μπορέσουν να μας τα παρουσιάσουν. Από μόνοι θα ε, έρθουμε σε επαφή μαζί σας για τον προπολογισμό του 2020 αφού πήγε καλά η πρώτη φάση συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής μας και έχουμε και πρόεδρο στον οποίο επιστρέφω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μπόρεσα να σας παρουσιάσω σύντομα πώς έχει η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των οργανισμών. Έχουν περιορισμένο χρονικό διάστημα και γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να μιλήσετε έξι λεπτά ο καθένας, να το τηρήσετε αυτό. Η κυρία Μόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, καταρχάς συγχαρητήρια επί τη εκλογή σας ε, στη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Εύχομαι σε όλους σας κάθε επιτυχία στην θητεία σας, στην κοινοβουλευτική. Είμαι εδώ υπό την ιδιότητά μου σαν παρούσα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Οργανισμών. Και όπως είπε και ο πρόεδρός σας στην αρχή, θα ήθελα να παρουσιάσω το δίκτυο σε εσά, να σας εξηγήσω λίγο πολύ ε, τι κάνουμε, ποιοι είμαστε. Λοιπόν, το δίκτυο έχει 45 μέλη και εκεί συμπεριλαμβάνουμε αποκεντρωμένες υπηρεσίες ως επιτοπλίστων, κοινοπραξίες ε, και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για παραδείγματος χάρη τεχνολογία. Έχουμε και άλλους φορείς που συμμετέχουν. Όλοι αυτοί οι φορείς και οι υπηρεσίες είναι ξεχωριστές νομικές οντότητες και καλύπτονται τη δευτερογενή, συστήνονται από τη δευτερογενή νομοθεσία και έχουν ε, συγκεκριμένα καθήκοντα διοικητικά, τεχνικά, οργανωτικά και εφαρμόζουν πολιτικές της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό, παρόλο που μπαίνουμε στον πειρασμό να μας θεωρήσετε ότι είμαστε ένα, αλλά δεν επικρατεί μια ομοιογένεια στο δίκτυό μας. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τα μέλη των δικτών ανάλογα με πολιτικ... τομείς πολιτικής, ε, με διάφορες θεματικές, ε, θεματικές προσεγγίσεις, και καλυπτόμαστε από τι ειδικέ επιτροπέ του Κοινοβουλίου. Θα μπορούσαν να υποδιαιρεθούν και ανάλογα με το είδο των καθηκόντων που εκτελούν σε ρυθμιστικού φορεί που έχουν την εξουσία να υιοθετήσουν δεσμευτικού ε, κανόνε ή αποφάσει που έχουν άμεση συνέπεια όπω το θέμα, το γραφείο που είναι για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε και οργανισμού που παρέχουν τεχνική και επιστημονική γνωμοδότηση ή βάλουν εκθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη. Ο τελευταίος τρόπος να μας διακρίνεται είναι η δομή η χρηματοδοτική. Η κυρία Χολμάιερ ήδη αναφέρθηκε σε αυτό. Έχουμε πολύ ε, λίγους αυτοχρηματοδοτούμενους φορείς. Έχουμε κάποιους που μερικά αυτοχρηματοδοτούνται, όπως είναι η ΕΑΣΑ, και κάποιους φορείς που εν μέρει χρηματοδοτούνται από εθνικές αρχές, όπως η Τραπεζική Αρχή, και οι περισσότεροι από εμά εξαρτώμεθα απόλυτα από τους πόρους Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως η CTC ή η ΕΦΣΑ. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω γιατί έχουμε αυτό το δίκτυο κοστίζουμε κάτι, αλλά προσφέρουμε και κάποια αξία για αυτά τα χρήματα και το δίκτυο έχει επίγνωση της ανάγκης βελτιστοποίησης της χρήσης των πόρων ε, και για αυτό το λόγο θέλαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και συντονισμένα να αντιμετωπίζουμε πολιτικέ όπω ο κανονισμό, ο προσωπικό και δημοσιονομικό κανονισμό κλπ. Να συμμορφωθούμε με τι νέε νομοθεσίε και να ανταποκρινόμαστε και στι απαιτήσει για στοιχεία που μα ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί, οι θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και να έχουμε ενίο σημείο επαφή και εφαρμόζουμε τι δράσει τη κοινή προσέγγιση και βασικό στόχο είναι πραγματικά να αποφύγουμε επικαλύψει και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τα καθήκοντα κάθε οργανισμού. Παρέχουμε σε εσά τελικά ενίο σημείο επαφής και όχι 45. Προστιθέμενη αξία των οργανισμών. Όλοι μας μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα. Επέλεξα από τους οργανισμούς που ξέρω καλύτερα να σας παρουσιάσω Κάνουμε αξιολογήσει κινδύνου για νέου ε, κινδύνου από ε, μολυσματικέ ασθένειε και διάφορα κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει να μην το κάνουν από μόνο τους, μόνα του αυτά, αλλά έχουν διαθέσει πόρου ε, για ανάθεση άλλων καθηκόντων και εμεί κάνουμε τη δουλειά αυτή για τα κράτη-μέλη. Μετά έχουμε κάνουμε εποπτεία για τις μεταδοτικές ασθένειες, όπου το ECDC προηγουμένως είχαμε 17 διαφορετικά μέσα επίπεδα Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τώρα έχουμε ένα. Οπότε αυτοί οι πόροι διατίθενται ε, σε άλλα καθήκοντα. Λοιπόν, βρισκόμαστε 23 διαφορετικά κράτη-μέλη, αντιμετωπίζουμε συνεπώς προβλήματα που δεν αντιμετωπίζουν άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Για λόγους χρόνου να αναφερθώ στο συντελεστή, το διορθωτικό. Περί τίνος πρόκειται. Ε, είναι κάτι που επηρεάζει 21 από τους φορείς μας και και μειώνει την ελκυστικότητα του ε, οργανισμού σαν χώρο εργασίας. Δηλαδή, κάποιες υπηρεσίες παρέχουν τον ίδιο μισθό ε, θεωρητικά, αλλά στην πράξη η αμοιβή είναι 30% μικρότερη και αυτό οδηγεί και σε γεωγραφικές ανισορροπίες. Βλέπετε λοιπόν εδώ για κάποιους οργανισμούς κάποια παραδείγματα ε, είναι δύσκολο οι υπηρεσίες να ανταποκριθούν στις απαιτήσει που το άρθρο 27 του κανονισμού προσωπικού που απαιτεί γεωγραφική ισορροπία ε, στο μέτρο του δυνατού όσον αφορά το εργατικό δυναμικό η δυναμία να προσελκύσουμε επαρκή αριθμό ε, υποψηφίων με προσόντα ένα πρόβλημα. Και στις αιτήσει βλέπει κανείς ότι έχουν περιορισμένες αιτήσει, δύσκολο να κρατήσουμε το προσωπικό. Αν πάνε σε έναν οργανισμό θέλουν να βρουν θέση αλλού μετά. Ε, και στο τέλος αυτό έχει αντίκτυπο στην αποδοτικότητα ε, και κοστίζει. Η αναθεώρηση του διορθωτικού συντελεστή δεν προβλέπεται πριν από το 2023. Μέχρι τότε λοιπόν οι υπηρεσίες πρέπει να καλύψουν τα κενά μέσω κοινωνικών μέτρων που δεν είναι κάτι αποτελεσματικό, όπως καταλαβαίνετε. Εν κατακλείδη λοιπόν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, θα βρούμε νέες τρόπους συνεργασίες, οπότε ε, παρουσιάζουμε αυτή την πενταετή πρασιγική Έχουμε κοινή πύλη για τους διαγωνισμούς. Έχουμε εξοικονομήσει ήδη 10 εκατομμύρια ευρώ την πρώτη τετραετία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και ένα κομμάτι αυτών των οικονομιών ε, αφορά επίσης και την χρηματοδότηση. Ε, έχουμε κοινή υπηρεσία για τα απόκριση στις καταστροφές. Αυτό εξοικονομεί χρήματα. Προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας. Έχουμε κοινό στόχο. Αυτοί που μας χρηματοδοτούν, δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολίτες, θέλουμε να τελικά να βλέπουν κάποια αποτελέσματα τα χρήματα που μας δίνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ντεμπόλα. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εσείς κύριε Πρόεδρε και εσείς κυρία ε, εισηγήτρια, σας ευχαριστώ που επιτρέπετε στην Ευρωπόλ να παρουσιάσει την δημοσιονομική της κατάσταση. Λίγα λόγια πρώτα για το σημαντικό έργο της Ευρωπόλη μετά να μου επιτρέψετε να μιλήσω για τα αιτήματά μας για το προϋπολισμό του 2020. Η αποστολή μας είναι να υποστηρίζουμε τις χώρες μέλη στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος υπό όλες τις μορφές του, κυβερνοέγκλημα και τρομοκρατία. Δεν λαμβάνουμε κατασταλτικά μέτρα. Έχουμε περάσει από μια φάση διαρκούς ανάπτυξης και είμαστε πλέον ένας αξιόπιστος εταίρος όλων των δυνάμεων επιβολής του νόμου στις χώρες μέλη ο οργανισμός μας είναι ε, σεβαστός, στρατηγικός εταίρος, προσφέρει expert input στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκολύνει τις ε, διαβουλεύσεις στις ομάδες εργασίας και βεβαίως προσφέρει στήριξη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της τρομοκρατίας, σας θυμίζω τις εκθέσεις μας για την αξιολόγηση του κινδύνου που αποτελούν τη βάση για την ε, ε, κατάσταση των ε, πολιτικών. Επίσης, επιχειρησιακή στήριξη προς τις εθνικές αρχές που είναι βασικός στόχος των δράσεων της Ευρωπόλ. Προσφέρουμε και τα αναγκαία εργαλεία και την υποστήριξη πληροφορίες για εγκληματικές οργανώσεις, για τρομοκρατικές οργανώσεις. Έχουμε μια πολύ ασφαλή βάση δεδομένων, μπορούμε να διασυνδέσουμε τις χώρες μέλη προβαίνουμε σε εγκληματολογικές αναλύσεις, οι οποίες βοηθούν πλέον τους ερευνητές των χωρών μελών στο έργο τους. Από το 2015 εμπλεκόμεθα βαθιά σε όλες τις έρευνες επιθέσεων κατά της Ευρώπης και θυμίζω το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Στοκχόλμη, τη Βαρκελόνη, βεβαίω σε συνεργασία με την Eurojust και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Δικανικής Συνεργασίας έχουμε 240 αξιωματούχους συνδέσμους από 50 χώρες. Αυτό είναι κάτι το μοναδικό σε όλο τον κόσμο και διευκολύνει την καθημερινή συνεργασία μεταξύ εταίρων που έχουν εμπιστοσύνη οι στους δε. Είναι πολύ σημαντική η εργασία αυτή. Επίσης και η ε, ιατροδικαστική εργασία και στην Μάλτα μετά από τον ε, φόνο της Ντάφνη ε, Καρουάνα, αλλά και στην Σλοβακία μετά από τον φόνο του δημοσιογράφου εκεί. Υπάρχει διαρκής αύξηση ε, της ζήτησης των υπηρεσιών μας. Λαμβάνουμε σήμερα τετραπλάσια μηνύματα σε σύγκριση με το 2010. Πέρσι μόνο 1,1 εκατομμύρια μηνύματα η αδίποτε επένδυση στην Ευρωπόλ είναι επένδυση προς το καλό, υποφελία δηλαδή των χωρών μελών. Να εξηγήσω τώρα τις ανησυχίες μας σχετικά με την πρόταση για τον προϋπολισμό 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Δεκέμβριο του 2018 το Διοικητικό μας Συμβούλιο κατέθεσε σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 174,8 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί στο διοικητικό αυτό συμβούλιο εκπροσωπούνται οι χώρε μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά τα μέλη θεώρησαν ότι αυτή η αύξηση ήταν απολύτω δικαιολογημένη λόγω τη αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών τη Ευρωπόλ. Δυστυχώ. Στο σχέδιο 2020, του 2020 υπάρχει κενό 33,7 εκατομμυρίων και 32 θέσεων του οργανογράμματος. Η Ευρωπόλ έχει ωστόσο ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για το 2020, διότι ανταποκρινόμαστε σε άμεσες ανάγκες των χωρών, άμεσες επιχειρησιακές ανάγκες των χωρών μελών, όπως μας εξηγούν οι επικεφαλεί των αστυνομιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και σα φέρνω μερικέ προτεραιότητες. Ανάπτυξη της, ε, της ε, πλατφόρμας κρυπτογράφησης, ε, αντιμετώπιση της σωματεμπορίας, αντιτρομοκρατία, για την αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού από το διαδίκτυο, αντιμετώπιση ακραίων ε, βίων πράξεων που προέρχονται από την άκρα δεξιά, παρεμβάσεις σε κρίσεις ε, τρομοκρατίας, η ανάπτυξη του σχετικού κέντρου, διότι μόνο 2% από τα ε, κέρδη από το έγκλημα ε, δημεύονται στην ε, Ευρώπη. Μόνο 2% και βεβαίω και εγκλήματα κάτω του περιβάλλοντο. Θα μπορούσα να συνεχίσω. Θα αντιμετωπίσουμε μάλιστα πολύ δυσχερεί προκλήσει στο μέλλον, αν δεν έχουμε επαρκή χρηματοδότηση. Ο κύριο εταίρο μα είστε εσεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μα έχετε πολύ υποστηρίξει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Οι κατευθυντήριε γραμμέ για τον προπολογισμό του 2020 που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2019 προβλέπουν ρητά ενίσχυση τη Ευρωπόλ και τονίζουν την ανάγκη ενισχυμένη επένδυσης από πλευράς ευρωπαϊκής για την εσωτερική ασφάλεια. Επένδυση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων που δεν συμβαδίζει με αύξηση επενδύσεων για την εσωτερική ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, το κυβερνοέγκλημα είναι πολύ σημαντικές απειλές για την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και που χρειάζεται την απόλυτη προσοχή μας. Μπορείτε να είστε βέβαιε και βέβαιοι ότι κάθε δεκάρα που θα επενδύσετε στην Ευρωπόλ θα είναι εποφελία των κρατών μελών και των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κυρία Ντεμπόλερ. Ο κύριο Κι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Κυρία Συγήτρια, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, σας ευχαριστούμε που μας επιτρέπετε να προσέλθουμε και να παρουσιάσουμε την κατάσταση της ε, ΆΣΑ. Να αρχίσω με μία περιγραφή των καθηκόντων μας, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες. Κατά βάση έχουμε τέσσερα βασικά καθήκοντα. Το πρώτο είναι η σύνταξη της σχετικής νομοθεσίας για τις ε, για την αποστολή μας. Δεύτερο, να πιστοποιούμε όλα τα προϊόντα τα οποία, οτιδήποτε πετά δηλαδή στην Ευρώπη και τα ε, ε, αεροπλάνα Boeing δηλαδή τα οποία πετούν στον αέριο χώρο της Ευρώπης και όλες τις οργανώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες παγκόσμια σε ευρωπαϊκές αεροπορικές γραμμές. Δηλαδή, αν έχω μία πτήση KLM που πηγαίνει στο Μεξικό πρέπει να πιστοποιήσει η ΕΑΣΑ τους ε, παρόχους υπηρεσιών συντήρησης των αεροσκαφών τη ΚΑΕΛΕΜ στο Μεξικό. Επίσης, εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τέταρτο, προώθηση της χρήσης ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προτύπων, συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ώστε να επιτευχθεί το δυνατό επίπεδο ασφαλεία για τους Ευρωπαίου σε, ε, ε, σε όλο τον κόσμο. Αν εξετάσουμε τώρα τη χρηματοδότηση του οργανισμού μας, ΕΑΣΑ, εκεί διαφέρουμε λίγο από τους περισσότερους άλλους οργανισμούς με την έννοια ότι περίπου 60% ε, της χρηματοδότησής μας προέρχεται από τέλη της βιομηχανίας. Δηλαδή, όταν πιστοποιούμε ένα Boeing, λαμβάνουμε ένα τέλος, εισπράττουμε δηλαδή ένα τέλος από την εταιρεία Boeing ένα τρίτο περίπου από επιδοτήσεις, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και λαμβάνουμε επίσης και εισφορές από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν όμως αποφασίσει να είναι συνδεδεμένες χώρες της ΕΑΣΑ. Και το τελευταίο μέρος του, ε, ε του προϋπολογισμού μας πρόκειται για τα λεγόμενα earmarked funds ε, στο πλαίσιο δηλαδή της διεθνούς συνεργασίας για προγράμματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το χρηματοδοτικό μας μοντέλο δηλαδή είναι του ε, ειδικού δεσμευμένου εισοδήματος. Δηλαδή δεν μπορεί να μεταφερθεί αλλού το εισόδημα αυτό. Και για κάθε μια πηγή χρηματοδότησης έχει αυτή υπακούει στους δικούς τους κανόνες. Δηλαδή Εάν δεν καταναλωθούν όλα τα χρήματα που προέρχονται από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, οφείλουμε να τα επιστρέψουμε. Ή, εάν ξεπεράσουμε το όριο, πρέπει να αφαιρεθούν τα χρήματα που έχουμε ε, καταναλώσει παραπάνω από τον επόμενο προϋπολογισμό. Άρα το σύστημά μας είναι απολύτως στεγανό, είναι απολύτως στεγανά τα διάφορα δοχεία τη χρηματοδότησή μα μεταξύ του. Τώρα θα σα πω λίγα λόγια για το ποιε είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε σχετικά με τι πηγέ χρηματοδότηση. Το πρώτο, δηλαδή τέλη και χρεώσει. Εκεί έχουμε μια αγορά η οποία αναπτύσσεται ταχύτατα και τα τέλη και οι εισφορέ μα, ε, ωστόσο, ε, καθορίζονται μέσω επιτροπολογία ανά πενταετία. Έχουμε φτάσει τώρα πια σε ένα στάδιο όπου δεν ε, είμαστε συγχρονισμένοι πλέον με τις αγορές που εξυπηρετούμε και αυτό ισχύει ιδίως, μάλλον αυτό οδηγεί σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την καινοτομία στην, ε, ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Θέλουμε να αρχίσουμε δηλαδή να συνεργαζόμαστε με κάποιους οργανισμούς ή εταιρείες, αλλά δεν έχουμε την κατάλληλη ε, δομή τελών και έτσι αποφασίζουν αυτές οι επιχειρήσεις να πάνε στην Ιαπωνία ή στην Κορέα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αξίζει να μνημονεύσω επίσης από τη δική μας πλευρά ότι ο οργανισμός ΕΑΣΑ είναι ο μοναδικός τέτοιος οργανισμός σε όλο τον κόσμο που δεν χρηματοδοτείται από τέλη που πληρώνει οι επιβάτες ή τέλη προσγείωσης απογείωσης ή τέλη στα κάψιμα η συμβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι το τμήμα του προπολογισμού που έρχεται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό έχει παραμείνει ίδιο τα τελευταία 5-10 χρόνια. Ενώ, ιδίω από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, ο ρόλο μα έχει ενισχυθεί. Και μάλιστα σημαντικά και διευρυνθεί. Κάτι το οποίο οδηγεί σε απόκληση ανάμεσα στα καθήκοντα που καλούμαστε να επιτελέσουμε και στους πόρους που διαθέτουμε. Τέλος, για τα earmarked funds, εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε με τέσσερι διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κάθε μια από τι οποίε έχει δικού τη κανόνε για τα χρηματοδοτικά τη εργαλεία. Κάτι το οποίο οδηγεί σε μεγάλη γραφειοκρατική επιβάρυνση, γιατί κάθε μια από τι γενικέ διευθύνσει έχει ξεχωριστέ, όπω είπα, διαδικασίε, κανόνε, δεν είναι ενοποιημένοι. Το δεύτερο, επίσης πρόβλημα είναι ότι λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να ανακτήσουμε πλήρως τα κόστη μας όταν εκτελούμε τα προγράμματα αυτά για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας εμποδίζει να επιτελέσουμε πλήρως το έργο μας. Ε, συνοπτικά εν τέλει, οι τρεις πηγές χρηματοδοτήσεως αποτελούν και σημαντικές προκλήσεις. Είναι όμως ε, ε απολύτως ειδικέ, ε, για την ΕΑΣΑ και για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει αυτές θα χρειαστούμε την συνεργασία και την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρο. Επιθυμεί κανείς να λάβει το λόγο για να θέσει ερωτήσεις ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά διαπιστώσατε ότι ο νέος μόνιμος εισηγητής για τους οργανισμούς δεν έχει ακόμα οριστεί. Είχα την τιμή να διατελέσω εισηγητής αυτό στην περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο, οπότε γνωρίζω ε, πολύ καλά ακόμα τα διάφορα προβλήματα και δυσκολίες χρηματοδοτικές ε, που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Ανέκαθαν έλεγα εγώ στην Επιτροπή μας ότι είναι υποχρηματοδοτούμενος ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, γύρω στα 150 δισεκατομμύρια, λίγο πάνω, λίγο κάτω, η πολιτική να κάνεις για τα κράτη-μέλη όσο επιτρέπει αυτό το ποσό. Και αυτό το διαπιστώνουμε ιδιαίτερα προετοιμάζοντας το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο όλο και πιο έντονα. Ότι δεν θα φτάσουμε τίποτα αυτά τα ποσά. Εάν οι επιπλέον υποχρεώσεις που επιβάλλουν τα ίδια τα κράτη-μέλη και χωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα οποία ε, επιφορτίζουν ε, να κάνουν τη βασική δουλειά τους οργανισμούς. Δεν πρόκειται να αρκέσει. δηλαδή εκχωρούν αυτές τις αρμοδιότητες, αλλά δεν είναι πρόθυμα τα κράτη-μέλη να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάζεται πολλές φορές ε, να λύσει αυτά τα προβλήματα και δεν τις λέω καθόλου γι' αυτό, εις βάρος των οργανισμών τους δίνει όλο και λιγότερα χρήματα από όσα αντικειμενικά χρειάζονται. Το βλέπουμε πάντα εδώ στην Επιτροπή μας ε, οργανισμοί που αναλαμβάνουν περισσότερες υποχρεώσεις, ε, κατά φυσικό τρόπο παίρνουν περισσότερα χρήματα, τα οποία όμως αφαιρούν από κάποιες άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή δεν φτάνει η κουβέρτα ποτέ. Ε, τραβάς το πάπλωμα και κρυώνει είτε τα πόδια και ζεστάνει το λαιμό, είτε το αντίθετο. Οπότε οξύνεται αυτή η υποχρηματοδότηση. Γιατί είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το μετακυλεί στου οργανισμού. Όπως είπε και η Μόνικα Χόλμαια, το είδαμε στου οργανισμού ασφαλείας, όπου έχουν αυξηθεί απαιτήσει ε, ε, και για το Frontex ας πούμε και τις άλλες προστασίες των συνόρων από πού παίρνουν τα λεφτά από την Ευρωπόλ μεταξύ άλλων. Και ως Γερμανοί πολιτικοί και άνδρες και γυναίκες ερχόμαστε αντιμέτωποι με την εξή κατάσταση. Ε, έρχονται οι Υπουργοί Ιστορικών των Κρατηδίων, επενούν την Ευρωπόλ και μας λένε κάντε κάτι γι' αυτό και εμείς τους στέλνουμε στους Εθνικούς Υπουργούς Οικονομικών, πηγαίνετε εκεί να τους τα εξηγήσετε. Για η υποστήριξή μας για τους οργανισμούς είναι δεδομένη. Αλλά το θέμα είναι τα κράτη-μέλη πόσο είναι πρόθυμα εκεί να ανταποκριθούν και να απελευθερώσουν κονδύλια. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο που οι οργανισμοί τα τελευταία χρόνια υπέφεραν ιδιαίτερα λόγω του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σύνολο προσωπικού όπου εκεί συγκέντρωσε το οργανόγραμμα όλων τον οργανισμό. Και υπάρχουν κάποιες ε, μεταφορές εκεί προσωπικού. Ε, σε κάποιο βαθμό γίνεται αυτό, αλλά κάπου βρίσκει και τα όρια του και επηρεάζει σοβαρά, ε, θέτει ένα αμφιβόλο τη λειτουργία την ίδια των οργανισμών. Και στο τέλος των διαπραγματεύσεων του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, μήπως θα μπορούσαμε να δώσουμε κάτι στα κράτη-μέλη. Ε, από εκεί, δηλαδή τα κράτη-μέλη που δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν, μπορεί να χρειαστούν να χρηματοδοτήσουν περισσότερο, αλλά μετά να έχουν αποκομίσει και μια νίκη, ας πούμε, γιατί θα πούνε ότι αυτό το γραφειοκρατικό τέρας που έχει δημιουργηθεί κάπως περιορίζεται. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, και εδώ στο Κοινοβούλιο, ε, ε, ε, είχαμε μείωση του προσωπικού κατά 5% παντού, επώδυνη, αλλά για ορισμένους οργανισμούς αυτή τη στιγμή αυτό απειλεί την ίδια του την ύπαρξη. Ε, χρειαζόμαστε δηλαδή λίγο περισσότερη προσοχή, λίγο περισσότερη καλή βούληση για τους οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνω λίγο κακός. Θα πρέπει να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι δικοί του οργανισμοί, ιδιαίτερα εκτελεστικοί οργανισμοί, δεν θα πρέπει να ε, πλήττονται από αυτή την ε, κούρσα εξοικονόμησης. Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τη χρηματοδότηση την αυτοχρηματοδότηση μάλλον των οργανισμών που θα πρέπει να ορθοποθήσει Σωστά είπε η Μόνικα Χολμάιερ ότι ε, τα δημόσια καθήκοντα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από το δημόσιο για να μην έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Υπάρχουν όμως κάποιες εμπορικές ε, δραστηριότητες που έχουν αυτοί οι οργανισμοί και μπορούν να πληρώνουν όσοι υποφελούνται αυτών των υπηρεσιών. Έχουμε προχωρήσει μένα, υπάρχει ακόμα δυναμικό ανεκμετάλλευτο και θα αγωνιστώ και στην επόμενη, την τρέχουσα δηλαδή γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντρέσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις που αφορούν τους οργανισμούς. Δεν αφορά μόνο τις, τους οργανισμούς που εκπροσωπείτε εσείς, αλλά και τους άλλους. Με το Brexit σχετίζεται η πρώτη ερώτηση δύο υπηρεσίες έπρεπε να μετακομίσουν λόγω του ενδεχομένου του Brexit από Λονδίνο στο Άμστερνταμ και στο Παρίσι νομίζω. Ερώτηση. Η διαδικασία πώς πάει. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα όσον αφορά την μετακίνηση των οργανισμών από Λονδίνο στο Άμστερνταμ και στο Παρίσι. Ξέρω ότι Υπήρξαν κάποια προβλήματα με τις συμβάσεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Η άλλη ερώτηση για τη Frontex. Ακούσαμε τι είπε η κυρία Βόντερ την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο είπε από χίλια, χίλια μέλη προσωπικό η Frontex θα πάει στα 10.000. Συζητείται επί το θέμα αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο η πρόταση που ακούσαμε. Θα ήθελα περισσότερα να ακούσω πάνω σε αυτό. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που σχετίζεται με αυτό. Υπάρχουν ίσως και θέματα διαχειριστικά στον αφορά την Frontex. Είναι μεγάλη διαφορά να έχει κανείς έναν οργανισμό με λιγότερους από χίλιους που εργάζονται για τον οργανισμό και μετά να μεγαλώσει και να έχει 10.000 μέλη προσωπικό, όπως είπε η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να ακούσω κάτι πάνω σε αυτό. Ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας με τη Frontex, μετά τις διακοπές. Μήπως όπως μπορείτε, όμως μπορείτε να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις τώρα πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Ζόνκερ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή η συζήτηση για τους οργανισμούς είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προσελκύει το ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτοί οι οργανισμοί δεν δημιουργήθηκαν για το τίποτα, εκτελούν όλοι οι οργανισμοί αυτοί το στόχο τους. Καμία φορά αναφέρονται οικονομικά προβλήματα, η έλλειψη χρηματοδότησης για κάποιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Εξού και η ερώτησή μου. Ίσως στην Επιτροπή Προπολογισμών μπορούμε να σκεφτούμε τον δεχόμενο δημιουργίας νέων οργανισμών. Είμαστε πάρα πολύ σημαντική επιτροπή και υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε ήδη για τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέους οργανισμούς. Έρχομαι στην ερώτηση που θέλω να θέσω λοιπόν τώρα τι γίνεται με τον οργανισμό για το άσυλο, την υπηρεσία το άσυλο. Από ό,τι θυμάμαι, το Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε την απαλλαγή για αυτό το φορέα. Και τον Οκτώβριο θα γίνει ψηφοφορία πάνω στο θέμα. Θα ήθελα να ξέρω τι συνέβη. Υπάρχουν ακόμα δράσεις που έχουν προγραμματιστεί Ξέρω ότι υπήρξαν προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών. Υπάρχουν προβλήματα διαφάνειας όσον αφορά την χρήση των πόρων στα πλαίσια αυτού του φορά. Ευχαριστώ. Ο κ. Κούς. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση έχω ή περισσότερες μιας. Στον εκπρόσωπο της ΕΑΣΑ ε, είπε προηγουμένως ότι ε, μέσα στα αεροσκάφη υπάρχουν και αεροσκάφη Boeing. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι για το 737. Ε, ε, αυτό το μοιραίο αεροσκάφος. Έχει εγκριθεί από την ΕΑΣΑ. Και αν ναι, έχετε εξετάσει μήπως ε, είχατε επιδείξει κάποια επιπολαιότητα ε, στη χορήγηση της άδεια. Το ίδιο ισχύει και στην Αμερική. Υπάρχει κίνδυνος τώρα να ε, αντιμετωπίσετε αξιώσεις για αποζημίωση που θα πρέπει να επομιστείτε εσείς στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Thank you, Madam. Σας ευχαριστώ, η κυρία Μάρκες. Ehm, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση που δεν αφορά ιδιαίτερα τους οργανισμούς, αλλά είναι κάτι που αναφέρθηκε από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών και την ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας έδωσε. του το διορθωτικό συντελεστή, τους διορθωτικούς συντελεστές θέλω να θέσω. Το θέμα αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους οργανισμούς. Είναι κάτι που αφορά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιπροσωπείες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημεία ε, ενημέρωσης και πληροφοριών στα διάφορα κάτι μέλη. Αυτός ο συντελεστής, οι συντελεστές ιδιορθωτικοί αφορούν όλους τους οργανισμούς, όλους τους θεσμούς, όχι μόνο τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Οργανισμών που έθεσε το θέμα αυτό και έθεσε το πλαίσιο των διαφόρων διορθωτικών συντελεστών. Όταν θα συζητήσουμε στο μέλλον το νέο κανονισμό για τους υπαλλήλους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, Ίσως θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και αυτό το ζήτημα, αλλά δεν θα είναι ένα θέμα που θα αφορά αποκλειστικά τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία εισηγήτρια, την κυρία Μόνικα Χόλμαε, για τη σαφέστατη παρουσίασή της για όλη ε, αυτή την περίληψη, τη σύνθεση της προηγούμενης εργασίας που μας παρουσίασε. Κύριε Πρόεδρε, μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες από τις παρουσιάσεις που είδαμε στις διαφάνειες, γιατί ήταν πολύ κατατοπιστικές και θα μας ενδιαφέρει. Θα ήθελα να αναφερθώ σε διάφορα θέματα. Συμμετέχω στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ, και τα θέματα ασύλου, καταπολέμηση τρομοκρατίας, πρόληψη εγκληματικότητας ε, με ενδιαφέρουν και με καθοδηγούν. Θα ήθελα να πω εδώ λοιπόν ότι έχω την αίσθηση ότι οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά έχουν πάρα πολύ επιχειρησιακές αρμοδιότητες ε, που φτάνουν μέχρι τη συγκεκριμένη δράση και αποστολή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια και πολύ πόρη. Ε, όπως ε, και ο συνάδελφος Αντρέζεν, θέλω να αναφερθώ κι εγώ στο Frontex και να ρωτήσω τι γίνεται εκεί με τη συνέπεια. 191 θα σας πω πολλούς αριθμούς. 191 ήταν οι θέσεις αυτές δημιουργήθηκαν το 2020. Ενώ ο ρυθμός που μας πρότεινε και παρουσίασε η κυρία Φόντερ Λάιεν να φτάσουμε στους 10.000 ε, το 2020 φύλακες, θα σήμαινε πάνω από 1.500 ετησίως. Δηλαδή ε, δεν έχουμε πάρει το σωστό δρόμο. Αυτό πώς δικαιολογείται. Ακόμα και αν είμαστε εντός του ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ήταν 700 με 800 επιπλέον συνοριοφύλακες και ε, λιμενικοί το χρόνο. Επίσης, εκπλήσουμε για ε, την περιορισμένη στελέχωση και τα μέσα που δίνονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αντίθεση με τις πολιτικές δηλώσεις και εξαγγελίες ε, για τη λειτουργία υπηρεσίας Γενικού Εισαγγελέα που θα οριστεί. Τρίτη ερώτηση για την Europol. Εγώ, ξέρετε, ζω στο Στρασβούργο. Εκεί δρεύει ένα κέντρο αστυνομική και τελωνιακή συνεργασία. Υπάρχουν πολλά στην Ευρώπη που συνεργάζεται στενά με την Europol και κάνει πάρα πολύ χρήσιμη δουλειά για την πρόληψη του διεθνούς εγκλήματος, του διασυνοριακού, για την ε, παρακολούθηση και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε πέρσι το Δεκέμβριο στο Στρασβουργό, ε, αναζητώντα αυτό το τρομοκράτη. Ε, γενικά, διασυνοριακή συνεργασία για τη σύλληψη των κακοποιών. Ε, σε αυτά τα θέματα είναι πολύ πιο ισχυροί οι εγκληματίες από τις εθνικές διοίκησεις. Άρα, χρειάζεται ευρύτερη συνεργασία στην Ευρώπη, ε, με την Europol και την Interpol που είναι διεθνής. Ε, και λοιπόν δεν κατανοώ καθόλου την ε, μείωση των πόρων. Επίση, θα ήθελα να ρωτήσω σαν τον συνάδελφο τι γίνεται με την υπηρεσία ασύλου. Γιατί και αυτό το εξήγηλε η κυρία Φόντερ Λάιεν, ότι νέε προτάσει, μάλλον σχετικά με τον νέο αυτό οργανισμό, αλλά έχω μπει στην ουσία των θεμάτων, ενώ εμείς είμαστε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, που περιοριζόμαστε στο να συζητούμε τα οικονομικά, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούμε και τις νέες ε, αρμοδιότητες που εχωρούνται και έχω και μια ε, έτσι, θέληση για αυτά τα θέματα και περιμένουν πολλά από εμά οι πολίτες. Θα πρέπει να βρούμε ρεαλιστικούς δρόμους στον προϋπολογισμό αλλά και αποτελεσματικούς. Και τέλος δεν μιλήσαμε για τη δική σας υπηρεσία, για το δικό σας οργανισμό κυρία Πρόεδρε του Δικτύου. Θα ήθελα όμως να πω ότι οι ασθένειε δεν γνωρίζουν σύνορα. Περνάνε τα σύνορα, δεν ζητούν θεώρηση διαβατηρίου. Και μακροπρόθεσμα είναι και αυτό ένα ζήτημα ε, πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστώ. Ορίστε. Σας ευχαριστώ. Μια σύντομη ερώτηση. Σαν τακτικό μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης, θα ήθελα λεπτομέρειες ή δυνατόν για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για θέματα εργασίας στην Πρατισλάβα. Θα έχει ενεργά και απαθητικά καθήκοντα. Πότε θα λειτουργεί πλήρως. Σας ευχαριστώ πολύ, διότι σαν ε, εκλεγής βουλευτής στο Ευρωκοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό να έχω λεπτομερείς πληροφορίες για τις 45 αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ. Κατανοώ τα προβλήματα της υποχρηματοδότησης των φορέων αυτών και το πρόβλημα των διορθωτικών συντελεστών. Το ανέφεραν και συνάδελφοι πριν Ίσως να υπάρξει δυνατότητα να συζητήσουμε τους συντελεστές του διορθωτικούς μαζί με το γενικότερο πρόβλημα που αφορά τους Ευρωπαίους δημόσιους υπαλλήλους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ρέλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατος. Δεν θέλω να καταχραστώ του χρόνου σας. Ετέθησαν συγκεκριμένες ερωτήσεις για κάποιους οργανισμούς και υπηρεσίες. Ο κ. Αντρέασεν για τη μετακόμιση της υπηρεσίας φαρμάκων από Λονδίνο προς Άμστερνταμ. Ήταν πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Καταλήξαμε σε συμφωνία για υπενικίαση των γραφείων που είχαμε στο Λονδίνο πριν. Βρέθηκε νέος ε, ενοικιαστής. Θα υπάρχει κάποιο κόστος βέβαια, αλλά αυτό το κόστος θα παραμείνει εντός του πλαισίου που υπευλήθη σε αυτή την Επιτροπή αρχές του έτους για την EMEA ε, στα πλαίσια των κτηρίων. Καλά μαντάτα. Αρκετά μέλη έθεσαν ερώτηση για τα σχέδια προσλήψεων και το ρυθμό προσλήψεων των 10.000 συνοριοφυλάκων της Frontex. Συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου επετέφθη από αυτού αρχές του έτους για το ρυθμό των προσλήψεων. Η συμφωνία προβλέπει οι 10.000 να προσληφθούν μέχρι το τέλος του 2027 μετά από ένα πρώτο μετριοπαθές βήμα αυτό το έτος, το πρώτο σημαντικό βήμα προσλήψεων θα γίνει του χρόνου. Προβλέπεται το σχέδιο προπολογισμού του 2020, το τέλος του 2020 θα πρέπει να έχουμε χίλιους μεθοριοφύλακες που θα προσληφθούν. Αυτό είναι σημαντικό πρώτο βήμα. Είπε η νεοεκλεγής ο πρόεδρος ότι θεωρεί ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να επιταχυνθεί, να ολοκληρωθεί το 2024. Ουδέν σχόλιο από αυτού σήμερα. Σίγουρα όμως θα το προσεγγίσει με το σωστό τρόπο και αν αυτό ισχύσει βέβαια θα επανέλθουμε σε αυτή την Επιτροπή την κατάλληλη στιγμή. Αυτό θα έχει σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες. Αυτό ξυπακούεται. Ο κ. Ζωνσάλ άλλη ερώτηση για τη διαδικασία δημιουργίας νέων οργανισμών και ότι αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να γνωμοτήσει επ' αυτού Πράγματι, αυτό προβλέπεται στη Διοργανική Συμφωνία. Στο σημείο 31 μάλιστα της Συμφωνίας προβλέπεται η επίσημη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο στη διαδικασία. Για να ολοκληρώσω, διότι ακούστηκε κάποια συγκεκριμένη επίκριση και από τις υπηρεσίες και από το Γενική Συγήτρια για τον προπολογισμό της Europol, πιστεύω ότι πρέπει να υπερασπιστώ τη θέση μας πάνω σε αυτό. Λάβαμε πλήρως υπόψη όλες οι σημαντικές ενισχύσεις που έλαβε τελευταία χρόνια η Europol. Ελήφθησαν όλα αυτά υπόψη και προσθέσαμε και την διόρθωση για τον πληθωρισμό. Η εξολόγηση των δημοσιονομικών αρχών τα προηγούμενα χρόνια βασίστηκε και έγινε, ήταν η βάση μας και έγινε και η κατάλληλη διόρθωση για τον πληθωρισμό. Υπολογίζουμε το τέλος του 2020 η Europol θα έχει 178 θέσεις κενές, περισσότερες από αυτές που είχαν προγραμματιστεί μάλλον, στην αρχή του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό δικαιολογείται, δεν αμφισβητώ την αξία αυτού. Θέλω να πω ότι η Ευρωπόλ στηρίχθηκε πολύ και από τα τρία θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία του προπολογισμού. Άκουσα προσεκτικότατα την κυρία Χολμάιερ. Από ό,τι κατάλαβα δεν παίρνει πολύ σοβαρά την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να επανέλθουμε από αυτού ε, τους επόμενους ε, μήνες. Ίσως θα πρέπει να σταματήσω εδώ και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πάμε πίσω στους οργανισμούς τώρα για απαντήσεις. Παρακαλώ όμως να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για να μην μας τελειώσει ο χρόνος. Κύριε Ερμάν, ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις που θέσατε. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας. Κάποιες ερωτήσεις ήδη εκαλύφθηκαν από το συνάδελφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την EMA, την Υπηρεσία Φαρμάκων και η ΆΣΑ δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, δεν θέλω να επισέλθω εδώ σε λεπτομέρειες. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως. Να ζητήσουμε να, κάνουν, να δώσουν απαντήσεις οι υπηρεσίες της ερωτήσεις σας. Θα έχετε από την πηγή την απάντηση, έτσι. Καλύτερο αυτό παρά οι πληροφορίε που μπορώ να σας δώσω εγώ σήμερα εδώ, αν συμφωνείτε. Έχουμε συνάδελφο της Frontex εδώ, που μπορεί να απαντήσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες που δεν καλύφθηκαν από τον συνάδελφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρχε μια ερώτηση που αφορούσε τον διορθωτικό συντελεστή. Ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα, όχι μόνο για τους οργανισμούς και υπηρεσίες. Γιατί είναι πρόβλημα για τους οργανισμούς. Είναι διότι είμαστε σε 23 χώρες και αντιπροσωπείες ε, των θεσμικών οργάνων έχουν παρόμοιο πρόβλημα γνωρίζουμε ότι η συζήτηση για τον συντελεστή δεν είναι κάτι πανεύκολο ε, επειδή είναι στο ίδιο τμήμα του προϋπολογισμού οι οργανισμοί. Εάν δώσετε κάτι σε έναν ε, οργανισμό, πρέπει να φέρετε κάτι από άλλο οργανισμό. Η συζήτηση δεν πρέπει να αφορά τη μείωση του διθωτικού συντελεστή για κάποιους οργανισμούς και υπηρεσίες. Υφίσταται για κάποιο λόγο ο συντελεστή. Δεν πρόκειται περί αυτού. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι οι οργανισμοί που τώρα έχουν χαμηλότερο συντελεστή να μπορέσουν τελικά να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι εύκολο όμως. Μπορείτε να έχετε αντίγραφα των παρουσιάσεων όλοι. Έχουμε αφήσει αντίγραφα. Τα έχετε για το νέο οργανισμό, για την εργασία, την απασχόληση, είναι κάτι καινούριο, θα κάνουμε το ίδιο εκεί, όπως για ΕΑΣΟ και ΕΜΑ ή EMEA, θα σας δώσουμε γραπτός κάποιες πληροφορίες για να διαβάσετε τις πληροφορίες με την ησυχία σας. Ε, πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Συνάδελφος ίσως από τη Frontex να πει κάτι εν συντομία. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, όπως ήδη ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νομοθετική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αναμένουμε ο κανονισμός να τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, αν του έτους. Οι οργανισμοί, ο δικορισμός μας και τα ενεχόμενα μέρη και φορείς, ε, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή για να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε την πολύ διευρυμένη εντολή ποιοι είναι οι φορείς, ε, είναι ο Frontex, ε, η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοροφιακή και όλοι οι αρμόδιοι φορείς και αρχές στα κράτη-μέλη που καλούνται να ε, συνυλοποιήσουν και να εκτελέσουν αυτά τα καθήκοντα. Δεν είναι μόνο δικό μας μέλημα. Ρωτήσατε για τη στελέχωση και, και τη χρηματοδότηση. Ξέρετε ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο μέχρι το 2027 από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το 2024 έχουμε την ενδιάμεση μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση και αναθεώρηση που αναμένεται να ε, γίνει. Άκουσα κάποιες δηλώσεις εδώ και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ε, κάτι για το προσωπικό. Τους 10.000, δεν θα είναι 10.000 υπάλληλοι αυτοί ε, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προσωπικού. Ορισμένοι θα είναι δικοί μας υπάλληλοι μέχρι 3.000. Οι υπόλοιποι 7.000 θα απαρτίζονται από ε, μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα αποσπασμένους μακροχρόνια ή βραχυχρόνια καλύτερα αποσπασμένους ε, από τις αρχές των κρατών μελών. Είναι μεικτό το οργανόγραμμα. Ε, όπως ακούσαμε, ο διορθωτικός συντελεστής επηρεάζει και το Frontex και ε, φοβούμεθα ότι θα έχει επιπτώσεις στη διαδικασία πρόσληψης των 3.000 γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό η έδρα των εργαζομένων είναι η Βαρσοβία. Και είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε και πιο διαρθρωμένο διάλογο ε, στην Επιτροπή σας, αν μας προσκαλέσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Κυρία Μπόλε. Thank you, Mr. I would like to thank... Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους και όλους για την υποστήριξη και την αναγνώριση του ρόλου της Ευρωπόλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για του 178 παραπάνω θέσει διότι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε ανάγκε λόγω μεταναστευτικού. Επίση για το κέντρο Αντιτρομοκρατία λόγω των επιθέσεων. Είχαμε και την Internal Referral Unit για την αφαίρεση παράνομου από το διαδίκτυο. Δεν μπορεί κανεί πλέον να συγκρίνει τη σημερινή Ευρωπόλ με το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν ο οργανισμό αυτό πριν 7 ή 8 χρόνια. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει ως συνέπεια ότι θα πρέπει να ανατρέψουμε τις προτεραιότητες μας και οι νέες προτεραιότητες θα πρέπει ε, να ε, εγκριθούν σε τομείς πάρα πολύ μεγάλη σημασία ε, για τις χώρες μέλη. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αφαίρεση Παράνομου Υλικού από το Διαδίκτυο για το πολιετές πλαίσιο θα έχει 20 εκατομμύρια και 6 εκατομμύρια του χρόνου. Εάν επιβληθεί τελικά αυτή η περικοπή, θα έχει συνέπειες για τις χώρες μέλη. Οι έρευνες ε, υψηλού επίπεδου και εκεί χρειαζόμαστε 5 εκατομμύρια τον χρόνο, ενώ έχουμε μόλις 3,5 και η υποστήριξη για την ΕΠΟ, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλαδή, δεν μπορούμε ακόμα να, αξιολο... να εκτιμήσουμε μάλλον το όγκο εργασία που μας περιμένει. Στον κανονισμό προβλέπεται ότι η Ευρωπόλ καλείται να υποβάλει αναλύσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για να μιλήσουμε τώρα και για τους συμβασιούχους ε, υπαλλήλου, όπως είπε η συγκήτρια σας κυρία Χόλμαιρ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μείωση του προσωπικού κατά 235 συμβασιούχους, από ναι, από 235 148 μέχρι το 2022. Πάρα πολύ σημαντική και απότομη μείωση του προσωπικού που θα ε, ε, επιφέρει ε, σημαντική αναστάτωση στις εργασίες της Ευρωπόλ. Εμείς έχουμε προβλέψει το προσωπικό αυτό σε συμφωνία με το Διοικητικό Συμβουλίο και μετά από διαβούλευση με τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών διότι άλλοι οργανισμοί επίσης προσλαμβάνουν ε, συμβασιούχους υπαλλήλους, για παράδειγμα για την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων και για διοικητική υποστήριξη. Όπως βλέπουμε τώρα έχουμε, η πρόταση λέει τρία χρόνια, αλλά ήδη το προσωπικό μας εγκαταλείπει, διότι βέβαια ο ιδιωτικός τομέας ε, τους απορροφά, ιδίως τους ε, ηλεκτρονικούς, ε, ε, ε, τους δηλαδή ηλεκτρονικών συστημάτων και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής εξεργασίας δεδομένων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απαντώ σύντομα στον κύριο Κούς που ρώτησε για την πιστοποίηση των Boeing. Θα μπορούσα να σας απαντώ επί πολλή ώρα, αλλά νομίζω δεν είναι αυτό το θέμα. Για την περίπτωση του, των Boeing οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι η ε, βασική αρχή πιστοποίηση και, να, για να μπορέσει το αεροσκάφο να πετάξει εδώ, πρέπει εμεί να ε, κυρώσουμε την πιστοποίησή του. Μετά από τα δύο ατυχήματα που συνέβησαν, έχουμε συνεργαστεί και με την ε, Boeing και με την Αμερικανική ε, Αρχή Πιστοποίησης για να πιστοποιήσουμε τις νέες αλλαγές που επιφέρονται στο ε, αεροσκάφος αυτό. Λόγω όλων αυτών και λόγω του γεγονότο ότι οι προσπάθειε πιστοποίησής μας συντονίζονται με τους Αμερικανούς αλλά και με άλλους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, ε, πιστεύω ότι δεν έχουμε φόβο από ε, αγωγές αποζημίωσης. Τέτοιες υπάρχουν κατά της Boeing βέβαια. Και το αεροσκάφος αυτό θα επανέλθει βέβαια σε ενεργό υπηρεσία μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές. Άρα δεν φοβούμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε αγωγές αποζημιώσεων. Τώρα, πριν δώσω πάλι το λόγο στην κυρία Χολμάιερ, έχω δύο πράγματα να πω εγώ. Πρώτα, οι παρουσιάσεις που παρακολουθήσατε σήμερα θα σας διανεμηθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και βέβαια και λόγω των συζητήσεων, μάλλον λόγω της φύσης των συζητήσεων, είναι σημαντικό να δούμε την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα είναι αυτό δυνατό. Θα οργανώσουμε λοιπόν ε, συνάντηση με εκπροσώπους της Νέας Επιτροπής το δυνατόν συντομότερο. κυρία Χόλμαερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείξατε. Οι οργανισμοί νομίζω χρειάζονται επίδειξη ενδιαφέροντος από το Κοινοβούλιο διότι οι οργανισμοί ε, συχνά θεωρούνται κάτι σαν πάρεργο και δεν αναγνωρίζεται απολύτω η σημασία τη δράση του γιατί δεν τη βλέπουμε καθημερινά και επιστώνουμε ακριβώ και καθημερινά πού βρίσκονται οι αιστείε των προβλημάτων. Επομένω, η στενή συνεργασία με του οργανισμού είναι αναγκαία. Καμιά φορά ακούμε τη μομφή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εμεί εδώ, η Επιτροπή είμαστε το μακρύ χέρι των οργανισμών. Αυτή τη μομφή εγώ την είχα θεωρήσει πάρα πολύ παράδοξη, διότι είπα ότι όταν αντιμετωπίζουμε τα θέματα των οργανισμών και θέτουμε αιτιολογημένα ερωτήματα και θεμητά ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο καθήκον μια επιτροπή Προπολογισμών. Διότι οφείλουμε και να ρωτούμε, που ίσω δαπανήθηκαν υπερβολικά πολλά χρήματα, που ενδεχομένω αλλού εν ώψη των αποστολών που αναλαμβάνουν οι οργανισμοί στη βάση των όσων έχει αποφασίσει Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, υπάρχει επαρκέ προσωπικό, υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση. Και βεβαίως διαπιστώνονται συχνά προβλήματα. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής και για την Ευρωπόλ, διότι τον αγώνα αυτό τον κάνουμε από καιρό. Στην εποχή της ε, εχμής των τρομοκρατικών δράσεων χρειάστηκε να προσληφθούν έξτρα πρόσωπα στην Ευρωπόλ, 85 ε, τον αριθμό, που θέλει τώρα να καταργήσει τις θέσεις αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημαντική λοιπόν μείωση του προσωπικού. Εάν τώρα για 28 χώρες μέλη και παραπάνω από 40 διαφορετικά είδη εγκλημάτων, οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία, για παράδειγμα γεννητήσια κακοποίηση παιδιών, τα οποία είναι πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από τα σύνορα και εκεί ε, απαιτείται συντονισμός δράσεων 37 χωρών συνολικά. Όταν μιλούμε λοιπόν για τέτοιες τάξεις μεγεθών, 500 άτομα προσωπικό, ε, τότε δεν είναι υπερβολικά. Αν δω τι προσωπικό διαθέτουμε στη Γερμανία, για παράδειγμα, θεωρώ ότι είναι απολύτως παράλογο να απαιτούνται τα πράγματα αυτά από την Ευρωπόλ. Και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει σωστά μία προσαρμογή. Αυτά μπορούν να γίνουν μέσα στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος, που δεν έγινε όμως. Άρα, σε ό,τι αφορά τι συστάσεις μα, όχι μόνο για το 2020 αλλά και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, πρέπει να εξετάσουμε τα πράγματα πολύ προσεκτικά, να δούμε πού ενδεχομένω χρειάζεται περισσότερα, πού ενδεχομένω δεν υπάρχει ανάγκη, αλλά και πού υπάρχουν ανάγκε διότι απειλούνται ανθρώπινε ζωέ και σημειώνονται σημαντικέ, βαρύτατε απειλέ στις επικράτειες των χωρών μελών μα. Τα είχαμε πει τότε και με την ΕΑΣΟΥ και ε, την ΕΑΣΑ μάλλον γιατί είχαμε πει θα πρέπει να συνεχίσουν να πετούν τα αεροπλάνα αυτά ή όχι. Είχαμε πει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουν να γίνουν σεβαστά τα πρότυπα που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συνεργασία και με τι άλλε συναρμόδιε επιτροπέ και γι' αυτό νομίζω πρέπει να παραμείνουμε, να παρακολουθούμε προσεκτικά το έργο των οργανισμών που είναι πολύ σημαντικό και βεβαίω που βασίζεται στο προγραμματισμό που κάνουμε εμεί για του οργανισμού. Και για το έτο 2020 λοιπόν αναμένω στενή συνεργασία. Ευχαριστώ για τις εισρωές που θα ε, φροντίσουν να θέσουν υπόψη μου οι ε, συνάδελφοί μου για την ε, ε, προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστώ, πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τους εκπροσώπους, τον οργανισμό και θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Proceed on our agenda. Προχωρούμε. Στην ημερήση σε στο σημείο 9 που αλλάξαμε χτες με το 17 και θα συζητήσουμε τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις για το 2019 και το 2020. Να θυμίσω στα μέλη ότι τα αποτέλεσματα του πρώτου γύρου εκτίμησης των πιλωτικών προγραμμάτων και των προπαρασκευαστικών δράσεων τα έχετε λάβει αρχές Ιουλίου. Θα παρακαλούσα τον κύριο Ιρέλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει το σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, όπως αναφέρατε, αρχές του έτους λάβαμε κατάλογο με 197 προτάσεις για προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλωτικά προγράμματα από το Ευρωκοινοβούλιο. Ήδη έχει γίνει αξιολόγηση αυτών. Σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει στο Κοινοβούλιο απάντηση στις 9 Ιουλίου έγκαιρα πριν από αυτή τη συνεδρίαση και από τον απογευματινό τριμερή διάλογο. Τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολογήσεως, και το υπογραμμίζω, επρόκειτο περί τεχνικής αξιολογήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πόρισμα ήταν ότι θεωρούμε από τις 197 προτάσεις, 34 προτάσεις ότι μπορούν να εφαρμοστούν ως, προτι... προτείνονται χωρίς αλλαγές, 38 προτάσεις θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με κάποιο ανασχεδιασμό της πρότασης των προτάσεων για τις υπόλοιπες οι 125 εναπομένουσες προτάσεις θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν ή δεν εφαρμόσιμες διότι είτε υφίσταται η δυναμική βάση είτε οι προτάσεις είναι παρόμοιες ή αλληλεπικαλύπτουν άλλες ε, πρωτοβουλίες. εξαιρετικά φέτος θα, γίνει δύο, θα γίνουν δύο γύροι αξιολόγησης. Αυτό οφείλεται, διότι τώρα έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο, είναι προφανές, τη δεύτερη ομάδα για αξιολόγηση τη λάβαμε αρχές του μήνα από τον εισηγητή. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είμαστε το μέσο της περίοδου των διακοπών, αλλά λάβαμε ήδη υπόψη μας το αίτημα μέχρι 5 Σεπτεμβρίου να σταλούν οι απαντήσεις, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμμορφωθούμε. Και έτσι να δώσουμε τη τεχνική αξιολόγηση όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα προτάσεων εν ευθέτω χρόνο. Αν χρειαστεί, και αν δεν είμαστε 100% έτοιμοι αυτή τη φορά, ίσως θα επεξεργαστούμε ομάδες, θα στείλουμε μια πρώτη ομάδα πριν τι 5 Σεπτεμβρίου και μια δεύτερη αμέσως μετά. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμμορφωθούμε με το χρονοδιάγραμμα και προσβλέπουμε και στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρέλ. Η κυρία Χολμάιερ, η Γενική Συγγήτρια, έχει το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το πρώτο γύρο αυτής της αξιολόγησης. Εξ όσων διαβλέπω, 4α34β 38, C28 και δ, 37. Ε, αυτό τι σημαίνει, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί ασφαλμένη την εφαρμογή, γιατί είτε ήδη καλύπτεται αυτό από τον προπολογισμό, είτε από άλλη στην νομοθεσία ή επειδή δεν εντάσσεται καθόλου στο νομικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά ε, τρόπος να εφαρμοστεί σωστά Παρακαλώ τους συναδέλφους να κοιτάξουν τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά προγράμματά τους για να δούμε εάν αυτά συνάδουν με τα όσα αποφαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πάντα τα εξετάζει πάρα πολύ σχολαστικά και τεκμηριωμένα. Είναι καλή η εκτίμηση και αξιολόγησή τους και στις περισσότερες περιπτώσεις αφετηρία για μας για τη λήψη των αποφάσεων. Το πρόβλημα είναι για μας ότι ε, ε, ο πρώτος γύρος έχει απορροφήσει όλα μας τα κονδύλια. Γι' αυτό παρακαλώ και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 5η Σεπτεμβρίου που θα ψηφίσουμε και λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες να το φροντίσει. Δηλαδή, οι συνάδελφοι, αν έρθουν οι προτάσεις στις 5 Σεπτεμβρίου, δεν θα έχουν τον χρόνο καν να αντιδράσουν. Θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον να δώσουν την ευκαιρία στους συναδέλφους να, απαντήσουν, να αντιδράσουν. Δηλαδή, στην αρχή της εβδομάδας εκείνης, στις 2 Σεπτεμβρίου, για να υπάρξει καν η ε, ευκαιρία να το μελετήσουν οι συνάδελφοι και να αντιδράσουν, να απευθυνθούν σε μένα από μη συγγήτρια και να το συζητήσουμε με τους σκιώδεις συζητητές. Ποια είναι τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις που θα υλοποιήσουμε και ποια θα είναι η τάξη μεγέθους. Δεν θα ήθελα εγώ να το αποφασίσω μοναχικά ε, ως ε, εισηγήτρια, αλλά θέλω να το συζητήσω με τους άλλους εισηγητές και τις άλλες πολιτικές ομάδες για να σας κάνω μία πρόταση ε, έτσι, που να στέκει στα πόδια της και να βρει και τη συνένεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το διάστημα των θερινών διακοπών και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παρακαλώ ως εισηγήτρια οι δικέ μας βάσεις ε, είναι το Α και το, το, Β, τα προγράμματα που έχουν μπει εκεί. Και παρακαλώ τις πολιτικές ομάδες να το ελέγξουν και να μου δηλώσουν εάν υπάρχουν και άλλες επιθυμίες. Ε, συναντηθούμε αρχές Σεπτεμβρίου για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, να το ε, κοιτάξουμε. Το 2019 είχαμε 75 νέα ε, πιλωτικά προγράμματα και ε, προπαρασκευαστικές δράσεις, 50 και 25 αντίστοιχα και η ίδια τάξη μεγέθους είναι και φέτος. Μας περιμένει λοιπόν αρχές Σεπτεμβρίου πολλή δουλειά ενδιαφέρουσα και συναρπαστική για να καταλήξουμε σε ένα πάνω κάτω λογικό κατάλογο για να μπορέσουμε όλοι να τον εγκρίνουμε ως βάση για τις διαπραγματεύσεις του προϋπολογισμού με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλος να σχολιάσει παρακαλώ. Εσείς. Uh, Είμαι ο κ. Λόου. Ήμουνα μέλος του κόμματος Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο και νέο μέλος της Επιτροπής Προπολογισμών. Γενικό σχόλιο, αν επιτρέπετε. Προβληματίζομαι σχετικά με την κατεύθυνση προς την οποία οδεύει η Ευρώπη και γιατί ανησυχώ, διότι εδώ συζητάμε για κεντρικά σχεδιασμένη κατανομή μεγάλων ποσών οικονομικών. Κάτι μοιάζει με τη Σοβιετική Ένωση που διένεμε από το κέντρο τα χρήματα και κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Και όπως είπα τα πράγματα και στα πλαίσια της Συμφωνίας Απόσης Βρετανίας ανησυχώ για τις υποκείμενες υποχρεώσεις που είναι πάνω από 200 δισεκατομμύρια. Στα πλαίσια της Επιτροπής Προπολογισμών έχω τεράστιες ανησυχίες ως σαν επιχειρηματίας Θεωρώ ότι εμείς σαν εδώ δεν μπορούμε να έχουμε το σωστό έλεγχο σχετικά με τη χρήση των χρημάτων του φορολογωμένου. Και αυτό μου δημιουργεί τεράστια ανησυχίε. Άκουσα σήμερα το πρωί τεράστια ποσά που διανέμονται και δεν αισθάνομαι άνετα. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να τα ελέγξουμε. Αυτό οδηγεί σε διαφθορά, σε στρέβλωση και δεν μπορεί να είναι σωστή λύση ούτε για αυτή την Επιτροπή ούτε για την Ευρώπη. Thank you. Mr. Ευχαριστώ. Κύριε Σόνκα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω διαφορετική άποψη, κάπως διαφορετική. Πιστεύω ότι τα πιλωτικά προγράμματα είναι πραγματική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν πρόκειται περί πρωτοβουλειών που προέρχονται από τη βάση. Είναι ένα νέο άνοιγμα που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς μέσω αυτών των πιλωτικών προγραμμάτων. Προφανώς χαίρομαι για το μεγάλο αριθμό αυτών και ενδιαφέρομαι κυρίως για τη δεύτερη σειρά που θα καταφτάσει, διότι υπάρχουν προγράμματα άκρως ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να μην κάνουμε διάκριση μεταξύ των προγραμμάτων που προέρχονται από την πρώτη ομάδα προτάσεων ή από τη δεύτερη. Να γίνει μια ιεράρχηση συναρτήση των προτεραιοτήτων ή των προβλημάτων που μπορούν να επιληθούν από τα πιλωτικά προγράμματα. Δεν θα πρέπει να δούμε πότε υπευλήθη το πρόγραμμα ή τι πόρους εκπροσωπεί. Ε, έτσι θα ήθελα να προσεγγίσουμε λοιπόν την επιλογή αυτών των προγραμμάτων που θελοποιηθούν. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα σχόλια, υπάρχουν ερωτήσεις. Η κυρία Χολμάιερ, ξανά το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ απολύτως και με το σχόλιο αυτό, διότι ουσιαστικά τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις είναι πρωτοβουλία από κάτω προς τα πάνω και όχι το αντίστροφο. Έρχονται από τις περιφέρειες συγκεκριμένες ή από τους βουλευτές που έχουν εκλεγεί δημοκρατικά. Δεν είναι κεντρικές υποδείξεις και οδηγίες από κάποιους. Είχαμε πολλά τέτοια πιλωτικά προγράμματα τα οποία άνοιξαν το δρόμο ε, για ε, πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε πολλούς τομείς. Και δεύτερον, μια που έχω τώρα την τιμή να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, θα έλεγα στους συναδέλφους ότι εμείς ελέγχουμε τον προϋπολογισμό, ε, αλλά αυτό δεν γίνεται εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, αλλά στην Επιτροπή Ελέγχου. Και αν έχετε δει πόσο αυστηρά και δρακόντια ελέγχουμε τον προϋπολογισμό, ε, θα ξέρετε τι γίνεται πραγματικά. Κοιτάξτε πώ δουλεύουν εκεί οι συνάδελφοι. Κάνουν πολύ καλή δουλειά στα πλαίσια τη επιτροπή. Εδώ όμω τα πιλωτικά προγράμματα και τι προπαρασκευαστικές δράσει. θα πρέπει εμεί να επιλέξουμε, ε, να αποφασίσουμε μάλλον ποια θα επιλέξουμε το Σεπτέμβριο σε μια επικοδομητική και φιλική ατμόσφαιρα και φυσικά ελέγχοντα και την ποιότητα των ε, έργων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν το έχει αυτό σαν ησυχία και μέλημα γιατί αν δεν είναι καλή ποιότητα δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ή να τα χρηματοδοτήσουμε από τον προπολογισμό, από το PDP. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και χαίρομαι και περιμένω με χαρά τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες παρεμβάσεις. Σύντομη παρέμβαση. Υποστηρίζω το αίτημα της κυρίας εισηγήτριας να γίνει η αξιολόγηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να γίνει το ταχύτερο δυνατόν, ούτως ώστε να συζητήσουμε τα αποτελέσματα των πιλωτικών προγραμμάτων και να υπογραμμίσω ότι αυτά τα προγράμματα είναι σημαντικά. Όχι μόνο διότι προτείνονται κάτωθεν από την τοπική αυτοδίκηση και από ενώσεις ερευνητών, είναι σημαντικά όμως διότι είναι πιλωτικά προγράμματα. Πιλωτικά, το υπογραμμίζω, άρα πειραματικά προγράμματα προτείνονται. Έχω υπογράψει πέντε προγράμματα εγώ. Ένα από αυτά αφορά τα big data και πώς να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της δημόσιας ε, διοίκησης εναντί των big data. Υπάρχουν και θέματα όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος. Υποστηρίζω τη χρηματοδότηση, τη διαφανή αυτών των προγραμμάτων ερευνητικών προγραμμάτων που θα είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τους πολίτες μας και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και βέβαια η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι σημαντικότατα στοιχεία, ύψιστη προτεραιότης, καμιά φορά όμως έχουμε και άλλα προβλήματα, τα ξέρετε. Μεγάλη γραφειοκρατία, γραφειοκρατικό έλεγχο, είναι πολύ σημαντικό αρχές Σεπτεμβρίου ή δυνατόν να έχουμε στα χέρια μας την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βίνζιχ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Τίποτα μονιμότερον της αλλαγής για τις περιφέρειες. <clears throat> Ε, είναι αναγκαίο να ληφθεί αυτό υπόψη. Όλοι σκέπτονται τώρα ενδεχόμενα καταχρήσεων και διαφθοράς. Ακούσαμε ήδη ότι η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού άλλωστε αυτό το ρόλο παίζει παρακολουθεί και ελέγχει. Πρέπει ίσως να σκεφτούμε αν ίσως ως νέες βουλευτές να δούμε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του Όλαφ, της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης των Απατών. Ευχαριστώ. Κύριε τις εσείς ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι είπατε επί της ουσίας για το μηχανισμό, τώρα έχω να πω τα εξής. Αυτή η μεθοδολογία πληρωμών ακριβώς έχει ως στόχο ε, να αποφεύγονται οι σπατάλες. Χρειάζεται λοιπόν να γίνεται ένα πρόγραμμα, ώστε ενδεχομένως να αποφευθεί να κατασπαταληθούν χρήματα στο μέλλον. Τα pilot project και οι προπαρασκευαστικές δράσεις ε, προετοιμάζονται μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η επόμενη Επιτροπή προβλέπει αρνητική αξιολόγηση. Εκεί είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Ε, γι' αυτό επαναλαμβάνω την έκκληση. Ελέγξτε εάν έχει γίνει η προπαρασκευή με έγκριση της Κομισιόν ή όχι. Θα μπορούσα να σας δώσω και παραδείγματα, έτσι. Ε, ευχαριστώ. Υπενθυμίζω σε όλους και όλους ότι το τμήμα πολιτικής Policy Department θα αναλύσει με λεπτομέρεια τα θέματα αυτά. Άρα θα μας δώσει ένα πλαίσιο για να μπορούμε να κρίνουμε και να βλέπουμε και πού πηγαίνουν τα χρήματα. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας ε, συνάντηση και επομένως ε, σας εύχομαι καλές διακοπές, καλές λιακάδες, αλλά θα χρειαστείτε και μάλλον και κάποιες σκίες. Επίσης, να αρχίσουμε αμέσως μόλις ε, αποχωρήσουν ε, τα μέλη μας με τους συντονιστές, γιατί νομίζω είναι και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να δράσουμε.